πιστώνεται η εγκυρότητα της εντολής της κυρίας ε, Κάρη. Οι αρμόδιες επιτροπές έχουν κάνει διορθώσεις για εννέα κείμενα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με το άρθρο 216, εδάφιο 4 του κανονισμού, θα θεωρηθούν εγκεκριμένε αυτές οι ε, διορθώσεις, εάν εντός 24 ώρου δεν διαφωνήσει μια πολιτική ομάδα τουλάχιστον 40 βουλευτές. Τα κείμενα θα